με σε ένα παρόμοιο ζήτημα. Και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ακολουθεί η δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής και υπάτου εκπροσώπου της Ένωσης ε, ε θέμα η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά την παράνομη εκλογή νέου Προέδρου και νέου Προεδρίου της Εθνοσυνέλευσης. Εάν συμφωνείτε... Δεν θα έχουμε κάτι αυτή τη φορά και η συζήτηση θα αρχίσει με την ομιλία και πάλι του είπα του εκπροσώπου. Κύριε Μπορέα, to... αν είστε έτοιμος. No problem, no problem. We are just completely okay. Thank you so much for ναι, μισό λεπτό, εντάξει, ευχαριστώ. For following this closely, thank you so much, High Representative. The floor is I was looking for the papers. Ψάχνω τα χαρτιά μου. An interesting debate. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και η τελευταία φορά τη Βενεζουέλα. A few weeks ago, this plenary... Πριν από λίγες εβδομάδες, συζητήθηκε εδώ στο Κοινοβούλιο η ανθρωπιστική ε, κρίση στη Βενεζουέλα μετά από το πολιτικό αδιέξοδο. Δυστυχώς σήμερα ε, θα συζητήσουμε την περαιτέρω επιδείνωση της πολιτικής κρίσης. Αυτό είναι αποτέλεσμα των εξωφρενικών υποθέσεων ε, κατά της δημοκρατικής λειτουργίας της Εθνοσυνέλευσης και την εκλογή παράνομου Προέδρου στη Βουλή χρησιμοποιήθηκε βία κατά του Προέδρου Γουαϊντό και πολλών βουλευτών στις 5 Ιανουαρίου για να μην εκλεγεί νόμιμα ε, η Εθνοσυνέλευση και το Προεδρείο της. δεν είναι μόνο μείζον επίθεση κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αλλά και περαιτέρω πόλωση της κατάστασης και κλιμάκωση η λεγόμενη εκλογή του Λουίς Μπάρβα δεν είναι νόμιμη, δεν σέβεται τις νόμιες διαδικασίες, ούτε τις δημοκρατικές ε, συνταγματικές αρχές, δεν υπήρχε απαραίτητη απαρτία, δεν υπήρξε πλειοψηφία και γενικά δεν έγινε ε, σεβαστός ο κανονισμός. Άρα δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τον νέο πρόεδρο της Βουλής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνής Ομάδα Επαφών γρήγορα αντέδρασε και τόνισε την υποστήριξη του Χουάν Γουαϊδό ε, ως ε, νόμιμου προέδρου ε, της Εθνοσυνέλευσης. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα, τα καταδικάζουμε και εκφράζουμε υποστήριξή μας στον κύριο Γουαϊδό χρειάζονται τώρα και άλλα περιοριστικά μέτρα απέναντι στους αρμόδιους που υπονομεύουν τη δημοκρατία. Βεβαίως τα μέτρα αυτά σε καμία περίπτωση δεν είναι εις βάρος του λαού της Βενεζουέλας που ήδη στενάζει. Στοχευμένες κυρώσεις ε, είναι ένα εργαλείο αλλά όχι το μοναδικό. Χρειαζόμαστε και άλλες οδούς ε, συμπληρωματικές και επικοδομητικές Ακόμα και αν φαίνεται το μέλλον ζωφερό και δεν υπάρχουν προοπτικές για ε, προσεχή λύση του πολιτικού αδιεξόδου, θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε να δημιουργούμε πολιτικό χώρο για διαπραγματεύσεις για μια βιώσιμη επίλυση της κρίσης και αυτό μπορεί να προέλθει μόνο από γνήσιες διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ των νόμιμων εκπροσώπων και με την νόμιμη οδό. Ε, όταν μιλούμε για αποκατάσταση των θεσμών, ε, πρόκειται κυρίως για την Εθνοσυνέλευση και το Ανώτατο Δικαστήριο. Χωρίς τους θεσμούς αυτούς δεν νοείται ελεύθερη νομοθετική διαδικασία, βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, ούτε βιώσιμη λύση για τη Βενεζουέλα. Επανειλημμένα έχουμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αφισθεί προσπαθειών για να συνεχίσει να βοηθάει μια γνήσια διαδικασία χωρίς αποκλεισμού προς τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου με ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές. Άλλη προσπάθεια είναι να έχουμε μια πιο συντονισμένη προσπάθεια προς την κρίση στη Βενεζουέλα από τη διεθνή κοινότητα. Θέλω να ζητήσω από τον ειδικό ε, σύμβουλο ε, Ιγκλέσιας και Ιγκλέσια. μην μπλέξουμε τώρα του Ιγκλέσια, μην γίνει καμία παρεξήγηση. Μιλώ για τον και Ιγκλέσιας. Ε, έτσι ώστε ε, να ε, υπάρξουν συντονισμένες διεθνείς προσπάθειες. Καταληκτικά θα έλεγα ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε επαφή με άλλους διεθνείς παράγοντες. Πάντως ένα είναι βεβαίω χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμό τη διεθνούς κοινότητα επιγόντως. Έτσι μπορώ να συνοψίσω αυτά που θέλω να σας πω και είμαι βέβαιος ότι και από τη συζήτηση ε, θα καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Το προεξοφλώ. Χρειαζόμαστε πιο συντονισμένες προσπάθειες όλης της διεθνού κοινότητας και μάλιστα επιγόντως. Ε, αυτό το αδιέξοδο δεν μπορεί να συνεχίζεται διαπαντός. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Θα αναζητήσουμε ισχυρή υποστήριξη από όλους τους ενεχόμενους παράγοντες και από την ομάδα επαφής. Θα ζητήσουμε να εξακολουθήσει τις προσπάθειές και τις εργασίες της. Η λεγόμενη διαδικασία του Όσλο έχει πίσω οδηγηθεί σε αδιέξοδο και τα δεινά και ο πόνος του λαού της Βενεζουέλας και η πολιτική κατάσταση απαιτούν να πιέσουμε περισσότερο για να γίνουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές όπως επανειλημμένα και εδώ και καιρό ζητούμε ανεπιτυχώς αλλά αυτά που έγιναν στην εκλογή του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης είναι καμπή και ορόσημο για μια κατάσταση που χρειάζεται τώρα μεγαλύτερη δέσμευση και δράση από πλευρά μα. Ελπίζω αυτό να γίνει τι επόμενε εβδομάδε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα αρχίζει η συζήτηση. από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Λόπες Χίλ. Ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση, έχοντας ακούσει την προηγούμενη, ε, με κάνει να σκέφτομαι ότι ε, και εδώ κάνουμε λίγα και πολύ καθυστερημένα. Ο Νικολά Μαδουρό προσπάθησε με στρατιωτική υποστήριξη να κάνει ένα εσωτερικό πραξικόπημα προκειμένου να απαγορεύσει ε, η Εθνοσυνέλευση να επιλέξει τον πρόεδρό της. Ε, ο στόχος ε, είναι να εμποδιστεί οποιαδήποτε προσπάθεια μετάβαση στη δημοκρατία. Το κοινοβούλιο μας μία ακόμα φορά θα πρέπει να εκφράσει την υποστήριξή του στον Χουάν Γουαϊντό όχι μόνο ως πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης αλλά και ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας. Το έχουν κάνει πάνω από 60 χώρες ε, και όργανα, παγκόσμια όργανα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ούτε τις αιτίε ε, ούτε τους αυτούργους ε, αυτού του πραξιοπήματος. Εξακολουθούμε να ζητούμε από τον είπα το να επιβληθούν κυρώσεις στους υπεύθυνους των κατάφορων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου. Ε, και οι Ρώσοι που να μην επηρεάζουν τον ίδιο τον πληθυσμό, αλλά τους, ε, ε, αυτούς που έχουν διαπράξει τις συγκεκριμένες πράξεις. Η χειρότερη κύρωση που μπορούμε να επιβάλλουμε στους πολίτες της χώρας αυτής είναι να μην δράσουμε για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Γιατί έτσι τους στερούμε το μέλλον τους. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Άλλος ένας κύριος Λόπες από τους σοσιαλιστές αυτή τη στιγμή. Όπως είπε ο υπατός εκπρόσωπος, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να καταγγείλουμε την απόπειρα ε, κοινοβουλευτικού πραξικοβήματος εκ μέρους της κυβέρνησης Μαδούρο. Το να παρεμποδιστεί η λειτουργία της ε, Δημοκρατικής Αθνοσύνελευσης της Βενεζουέλας ε, έχει ως ε, στόχο την αφαίρεση της ε, νομιμοποίησης που έχει η Εθνοσυνέλευση ε, και ο ίδιος ο Χουάν Γουαϊντό, ε, τον οποίο πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει ως προσωρινό πρόεδρο της χώρας. Να υπενθυμίσουμε ότι παίζουμε ένα επικοδομητικό ρόλο εμείς εδώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν τρόπο που ενδεχομένως απογοητεύει το καθεστώς το οποίο δεν βρίσκει ε, παράθυρο ευκαιρίας ε, δεν οδηγεί τη χώρα στην δημοκρατία. Ε, είμαστε υπέρ των ε, εστιασμένων κυρώσεων, αλλά ταυτόχρονα δρούμε και μέσω της ομάδας επαφής προκειμένου να γίνει ένας διάλογος που θα οδηγήσει σε ελεύθερες εκλογές. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κάνιας. Εκ μέρους του Renew Europe. Αυτό, το, αυτό δεν είναι απλώς μια συζήτηση, δεν πρέπει να οδηγεί σε μια ακόμα απλώς δήλωση. Με το ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει α, τα τεκτενόμενα στη Βραζιλία ε, και καταγγέλει το τυραννικό καθεστώ του Νικολά Μαδούρο για αυτό που ήταν μια απόπειρα κοινοβουλευτικού πραξικοπήματο παρεμπόδιση τη λειτουργία των δημοκρατικών δεσμών. Είναι μια φάρσα αυτό το καθεστώ και αυτό το πραξικόπημα το αποδεικνύει. Οι βουλευτέ αυτοί έχουν εκλεγεί δημοκρατικά και παρεμποδίζονται. Έχουμε αναγνωρίσει τον Χουάν Γουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο για την Εθνοσυνέλευση ως μοναδικό δημοκρατικό θεσμό στη χώρα. Πρέπει οι βουλευτές της να τη χάνουν σεβασμού και το καθεστώς δεν πρέπει να τους να ασκεί πίεση εναντίον τους. Ζητά το ψήφισμα ε, από τον το εκπρόσωπο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί των προσπαθειών να επανέλθει η δημοκρατία στην ε, Βενεζουέλα σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της Εθνοσυνέλευσης μέσω της ομάδας επαφής. Ζητούμε να ενισχυθούν οι κυρώσει σε αυτού που είναι υπεύθυνοι για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την καταστολή και την καταπίεση. Και ζητά το ψήφισμα αυτό από τα μέρη τα οποία δεν έχουν αναγνωρίσει τον Χουάγου ως ω προσωρινό πρόεδρο να το πράξουν. Ζητούμε από τους, και ζητούμε επίση οι πολιτικοί εκπρόσωποι τη Βενεζουέλα να αναγνωριστούν ω τέτοιοι. Το ψήφισμα τέλος απευθύνεται στον ίδιο το λαό της Βενεζουέλας ε, και απευθύνει ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα λέγοντάς του ότι δεν είναι μόνος του ο λαός. Μέσω μιας ευρείας πλειοψηφίας των εκπροσώπων του ο λαός αυτός ε, ζητάει από μας και θα το κάνουμε να σταθούμε στο πλευρό του, να ενισχύσουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις και την μετάβαση ε, σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ε, που θα δώσει ελπίδα. Ευχαριστώ. Κύριος Χάιτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι τραγική το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας, παραδείγματο χάρη, χαρακτηρίζει την κατάσταση ε, σε αυτή την χώρα που έχει τα περισσότερα πετρέλαια στον κόσμο. Ε, ε, λέει ότι υπάρχει αστάθεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ληστείες, βίες ληστείες, χρησιμοποιούνται πλαστικές σφαίρες, επίσης υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Αυτά είναι πολύ λυπηρά. Ε, όμως αυτό που όλοι αποσκεπούν είναι τα αίτια που έχουν οδηγήσει σε αυτό το χάος. Είναι ένας αριστερός δικτάτορας, ο οποίος ε, πραγματικά με κάθε μέσο παραμένει προσκολλημένος στην εξουσία ε, και θεωρεί ότι αν δεν τα καταφέρουμε με τις ψήφους θα τα καταφέρουμε με τα όπλα. Αυτό είναι το σύνθημα του Μαστού Μαντούρο. Ε, γι' αυτό λοιπόν το καθεστώς αυτό ε, αντιμετωπίζεται ως πρότυπο από πολλούς αριστερούς στην Ευρώπη. Ο αγώνας ε, κατά των βίων ακραίων είναι σημαντικός όχι μόνο στη Βενεζουέλα αλλά και στην Ευρώπη για να μην έχουμε και στην Ευρώπη καταστάσεις που υπάρχουν στη Βενεζουέλα. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Χέρμαν Τέρτς. Καλησπέρα σας. Μου αρέσει πολύ αυτή η αλλαγή ύφους που ακούμε εδώ και το είδαμε και στην μεγάλη συμφωνία που θα ε, έχουμε αύριο για να υπερψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα για τη Βενεζουέλα. Επιτέλους, ορισμένοι αποφάσισαν ότι θα πρέπει να ασκήσουμε μαζική πίεση στο εγκληματικό αυτό ε, καθεστώς των κομμουνιστών και των λαθρεμπόρων ναρκωτικών που ε, έχουν τη χώρα σε ομοιρία και τίποτα δεν τους ε, τρομάζει, όπως έδειξε αυτό το ε, θέμα της επίθεσης και ε, στην Εθνοσυνέλευση. Ο Μαδούρο και ο Παντρίνο και οι λοιποί δεν θα πρέπει να μπορέσουν να βγάλουν ένα δολάριο από τη Βενεζουέλα. Και κάνουν και επίδειξη πλούτου. Ε, ε, και ε, μάλιστα συνδέονται και με τους Ισπανούς κομμουνιστές που είναι και στην κυβέρνηση τώρα. Αλλά αυτά είναι ανισχυτικά Είναι κίνδυνος για την περιοχή. Ο Μαδούρο καθημερινά σκοτώνει τον πληθυσμό του και έχει ένα, μια ισχύ στη διαφθορά που έχει περάσει τον Ατλαντικό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πινέντα. Είναι παράξενο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει να στηρίξει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει ακόμα και την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης. Ε, ε, ε επέλεξαν τον κύριο Πάρα στη θέση του που είναι επίσης από την αντιπολίτευση. Ο κύριος Γκουαϊντό αντί να προσπαθήσει να μπει από την πόρτα κανονικά προσπάθησε σαν κατσίκι να πηδήξει ένα φράχτη. Ε, φάρσα δηλαδή και ξανά ε, αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος στην έδρα ενός περιοδικού. Μην ξεχνάμε ότι το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Έχει μανία με τις ε, αυτοανακηρύξεις. Ε, πέραν αυτού έχει βάλει στην τσέπη του ένα πολύ μεγάλο μέρος της βοήθειας που έχει σταλεί στη Βενεζου... στην ε, αντιπολίτευση της Βενεζουέλας. Ο... ο άνθρωπος αυτός ε, κατά βάση είναι νοσταλγός ε, της δικτατορίας, της ισπανικής δικτατορίας. δημιουργεί και στην Ευρώπη πράγματα φασιστικές τάσεις που νομίζαμε ότι είχαμε γλιτώσει. Ο κύριος ε, Ταγιάννη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα χαιρετούμε τους ε, βουλευτές από τη Βενεζουέλα, προασπιστές και αγωνιστές της δημοκρατίας στη χώρα του. Ο κύριος Γουαϊδό είναι εκλεγμένος πρόεδρος, δημοκρατικά πρόεδρος της Βουλής, απέναντι στις δυνάμεις του κυρίου Μαδούρου, του δικτάτορα προσπάθησαν διάφοροι στρατιωτικοί και λοιποί για άλλη μια φορά να σκοτώσουν ε, τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει τη δύναμη να αντιδράσει ε, και να μην ε, λέμε ότι όλα αυτά ε, αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη, μεγαλύτερο θάρρος εκ μέρους του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το Κοινοβούλιο είχε την αποφασιστικότητα πρώτο να αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας και θα το ξανακάνει υπερψηφίζοντας ένα έγγραφο που που είναι πολύ σημαντικό και όπου επιβεβαιώνεται ε, επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα αρνητικά που κάνει ο κύριος Μαδούρο εις βάρος του λαού του καταστρέφοντας τη δημοκρατία, καταπνίγοντας την ελευθερία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι σωστό να επιβληθούν κυρώσεις ε, εναντί όλων των υπευθύνων και αυτές οι κυρώσεις θα πρέπει να ε, επιβληθούν σε όλους αυτούς που έχουν παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και οικονομικά έπληξαν οικογένειες και πολλοί είναι οι ε, συνεργάτες του Μαδούρο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει όλοι μας να έχουμε το θάρρος να λάβουμε μια σκληρή στάση αποφασιστική απέναντι στον κύριο Μαδούρο και απέναντι στη δικτατορία της Βενεζουέλας. Ε, δεν πρέπει να παρετούμεθα από το να επιδεικνύουμε θάρρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Σάντος, ένα λεπτό τα όσα συνέβησαν στις 25 του μηνός στην Βενεζουέλα ε, οδήγησαν στην παρεμπόδιση των δημοκρατικών εκπροσώπων της ε, χώρας ε, να ασκήσουν ελεύθερα τη, τις λειτουργίες τους και τα καθήκοντά τους. Ξέπερασε το καθεστώς μια κόκκινη γραμμή και αυτό δεν πρέπει να γίνει δεκτό. Τέτοιου είδους γεγονότα χρησιμεύουν απλώς για να πολλώσουν ακόμα περισσότερο την κοινωνία στη Βενεζουέλα και να δυσχεράνουν τις προσπάθειες να αναζητηθεί μια πολιτική λύση. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται η κρίση ε, και η ταλαιπωρία του λαού της Βενεζουέλας ε, που ζει μια ανθρωπιστική κρίση ε, που αναγκάζει το 90% του πληθυσμού να ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Από την αρχή αυτής της κοινωνιστικής θητείας έχουμε κάνει τρεις συζητήσεις για τη Βενεζουέλα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα τελευταία δύο χρόνια το θέμα αυτό έχει συζητηθεί οκτώ φορές στην Ολομέλεια. Και αυτό το ψήφισμα είναι το έβδομο που εκδίδουμε για την Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Θα πρέπει από τα λόγια να περάσουμε στις πράξεις. Ο λαός της Βενεζουέλας έχει πια κουραστεί, δεν αντέχει έχει φτάσει στα ωριά του. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Επίτροπε, στηρίζω την αποφασιστικότητά σα στην εφαρμογή, στην επιβολή κυρώσεων που θα συνδέονται με αυτούς οι οποίοι παραβαίνουν τους δημοκρατικούς κανόνες ε, και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα. Ταυτόχρονα πράγματι θα πρέπει να συνεχιστεί η διαβούλευση μέσω της ομάδας επαφής προκειμένου να οδηγηθούμε σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές που θα τύχουν ε, τις παρακολούθησης από τη διεθνή κοινότητα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας διακόπτω, λέει η Πρόεδρος, αλλά ε, ξενυχτάνε και άλλοι συνάδελφοι. Η κυρία Τσαρζάνοβα για ένα λεπτό και σας ευχαριστώ που θα τηρήσετε το χρόνο σας, αν μπορείτε. Κύριε, ε, είπατε εκπρόσωποι, το 19 το τελειώσαμε με μια συζήτηση για τη Βενεζουέλα και το 2020 πάλι για τη Βενεζουέλα αρχίζουμε. Φανταστείτε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εμποδίζεται να μπει από την αστυνομία και να προσπαθεί να ε, ε, περάσει ένα φράχτη, να σκαρφαλώσει για να μπει στο κτίριο και στην αίθουσα. Ακούγεται παράλογο, αλλά αυτό συνέβη στη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο ε, της Βουλής Χουάν Γουαϊδό. Δυστυχώς αυτά πια δεν μας εκπλήσουν στην Βενεζουέλα. Όλο και περισσότερο φαίνεται ότι ο Μαδούρο δεν προτίθεται να αφήσει την εξουσία ούτε να διαπραγματευτεί μια πραγματική δημοκρατική μετάβαση. Η δημοκρατία θα έρθει μόνο όταν τον αναγκάσει η πίεση να διαπραγματευτεί τους όρους αποχώρησης της κυβέρνησή του. Επιμένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να πιέζει το καθεστώς με επιλεκτικές κυρώσεις και να τις διευρυνεί και στα μέλη των οικογενειών ε, των όσων υφίσταται τις κυρώσεις και ταυτόχρονα να υποστηρίζει το δημοκρατικό και ειρηνικό διάλογο. Η κυρία Περέιρα από την ΚΟΕ, παρακαλώ. Ναι. Έχουμε χάσει το μέτρημα των συζητήσεων εδώ για τη Βενεζουέλα. Σε κάθε συζήτηση αυξάνεται το τελείριο που τη χαρακτηρίζει. Ε, οι κυρώσεις ήδη υπάρχουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Βενεζουέλας και έχει, ε, αποτελούν θηλιά για την οικονομία της Βενεζουέλας αλλά και για τους ξένους και όπως τους Πορτογάλους που ζουν εκεί. Ε, ας μην ε, αγνοούμε, ας μην κρύβουμε ότι ο λαός εξακολουθεί να ανθίσταται και να διεκδικεί την κυριαρχία του ενάντια στις εξωτερικές παρεμβάσεις. Διεκδικεί το δικαίωμα να χτίσει ελεύθερα το μέλλον μιας χώρας που δεν θα γίνει ξανά απικία. Γι' αυτό το λόγο εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας μαζί τους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και τώρα επόμενος ομιλήτης, ομιλήτρια η κυρία Μοντέρο γία ε, Ένα λεπτό το καθεστώς ε, Μαδούρο έχει ε, παραβαίνει συνεχώς το σύνταγμα της Βενεζουέλας. Το πιο πρόσφατο επεισόδιο ε, οδήγησε στην ανακήρυξη, παράνομη ανακήρυξη του Λουίς Πάρα ως πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης παραβιάστηκαν μία ακόμα φορά οι αρχές της ε, δημοκρατίας χωρίς καμία εδώ, χωρίς καμία ντροπή. Το κοινοβούλιο μας το έχει πει ήδη και στο παρελθόν με προηγούμενα ψηφίσματα σε προηγούμενες συζητήσεις. Στηρίζει τον Χουάν Γουαϊντό και την ε, δημοκρατικά εκλεγμένη Εθνοσυνέλευση. Ε, ε, είμαστε αντίθετοι με το σφετερισμό της εξουσίας, καταγγέλουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποίε έχει προβεί ο Μαντούρο και το καθεστώ του και η συμμαχή του. Ε, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν οι απειλέ εναντίον των μελών της εθνοσυνέλευση. Λυπάμαι πάρα πολύ της, για την ε, προηγούμενη ε, συνάδελφο που είπε ότι ε, πρόκειται για εξωτερική παρέμβαση. Ας το πει αυτό στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει. Είναι αυτά τα λόγια της πορτογαλικής ε, αριστεράς που κλείνει συνεχώς τα μάτια σε μια αξιολύπητη κατάσταση μια κατάσταση που ντροπιάζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Ντάντι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, πριν από λίγε μόνο ημέρε, ακούσαμε για πολλωστή φορά ότι υπάρχει βία που ασκήθηκε από το Μαντούρο, ο οποίο ε, το καθεστώ του έχει καταδικάσει ε, σε πείνα ένα λαό που βρίσκεται σε μία από τι πιο πλούσιε περιοχέ του κόσμου. Τέσσερα στοιχεία, τέσσερα εκατομμύρια, εκατομμύρια είναι οι Βενεζουελάνοι που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. 11 είναι τα κιλά που έχουν χάσει κατά μέσο όρο όλοι οι Βενεζουάλοι. 85% ε, είναι το ποσοστό των φαρμάκων που δεν μπορούν να μπουν στη Βενεζουέλα ε, και 95% ε, έχει μειωθεί το ΑΕΠ με βάση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, πρεσβεύει τη δημοκρατία και την ελευθερία πρέπει μέσα από τη διπλωματία και μέσα από κυρώσεις να εξαναγκάσει το καθεστώς του Μαδούρο να παρετηθεί και να επισπεύσει τη διαδικασία προς δημοκρατικές εκλογές. Ένα μήνυμα το οποίο ε, δεν θα αφορά μόνο το καθεστώς της Βενεζουέλας αλλά και όλους εκείνους που τον στηρίζουν πάνω απ' όλα τη Ρωσία. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία Μπιλμπάο Μπαραντίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε. Μια βίαιη και ε, χονδροειδής απόπειρα ε, να βάλουν χέρι στη Βουλή και το καταδικάζουμε ε, στεναρά. Θυμηθείτε την ιστορία της χώρας. Θα πρέπει να στηρίξουμε τον Χουάν Γουαϊδό για να ξεπεραστεί η κρίση, να αναγνωρίσουμε τους εκπροσώπους του στο εξωτερικό, να στηρίξουμε μια ε, ερευνητική επιτροπή που θα εξετάσει την κατάσταση και να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ομάδα Επαφής για να βρεθεί η ειρηνική ε, λύση με ελεύθερες εκλογές με κυρώσει κατά προσώπων που έχουν παραβιάσει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Να φύγει από την εξουσία ο Μαδούρο γιατί τη Βενεζουέλα την έχει καταλήψει εδώ και χρόνια. Ε, είναι τεράστια η φτώχεια και τα δεινά που υφίσταται ο λαός και υποφέρει από τη δικτατορία του. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος ε, και τώρα το λόγο έχει ο, ο Αντιπρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε πέντε λεπτά αν θέλετε κύριε Μπορέ. Αν δεν έχετε κουραστεί πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας σήμερα. Uh, σας ε, πολλά από τα σχόλιά σας ε, δείχνουν ότι Ε, έχουμε διαφορετικές ερμηνείες σε γεγονότα όμως τα οποία έχουν, ε, ε, έχουν εκπέμφθει σε όλο τον κόσμο κατά την άποψή μου θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον Χουάν Γκουαϊντό ως πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης αυτό δεν πρόκειται από μόνο του να λύσει το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον αποτελεί μια κοινή θέση. Σημειώνω ότι το κοινοβούλιο είναι διχασμένο για το τι έχει συμβεί στη Βενεζουέλα, αλλά θα πρέπει να σταθούμε στα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι σαφή. Ο Χουάν Γουαϊδό είναι για μας ακόμα πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και κατά συνέπεια παραμένει και προσωρινός πρόεδρος της ε, χώρας ε, που καλεί σε εκλογές. Θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much for your... Ευχαριστώ πάρα πολύ, αξιότιμα μέλη. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος για την ολοκλήρωση της συζήτησης αυτής. Η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη. Ε, σας εύχομαι καλή χρονιά και καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ τον είπα εκπρόσωπο για αυτή τη νυχτερινή συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα. Αύριο το πρωί, Τετάρτη, 15 του μηνός, θα συνεδριάσουμε από τις 9 μέχρι τις 2 και ε, τις ε, ε, από τις 3 και μετά. Την ημερήσια διάταξη θα τη βρείτε στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Καλό σας βράδυ και πάλι. Καλή νύχτα σας.